Bonjour euh, tout le monde. J'ai le plaisir d'accueillir Madame le commissaire de l'action humanitaire qui est venue nous rendre compte. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Τζόρτζεβα, η οποία θα μας μιλήσει για την αποστολή της, τη σημαντική της αποστολή στο Πακιστάν και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον πρέσβη του Πακιστάν. Αυτό είναι και το μοναδικό σημείο στην ημερήσια διάταξη Υπάρχει κάποια αντίρρηση ή σχόλια επί του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Φαίνεται πως όχι, άρα εγκρίνεται η σχολια επι του σχεδιου ημερησια διαταξης φαινεται διάταξη. Το Πακιστάν επλήγει από την σοβαρότερη καταστροφή στην ιστορία του. Το ε, Πακιστάν επλήγει από πλημμύρες και άμεσα ή έμεσα έχουν πληγεί 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Το εύρος αυτών των πλημμυρών καταδεικνύει ότι θα πρέπει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ πολλές ε, περιοχές στο ε, βορειοδυτικό τμήμα της χώρας αντιμετωπίσουν δυσκολίες πρόσβασης και ασφάλειας. Για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την ε, κυρία Επίτροπο, την κυρία Τζόρτζεβα, η οποία μετέβη στο Πακιστάν και θα μας μιλήσει για τα αποτελέσματα της αποστολής της. Στη συνέχεια θα έχουμε μια σειρά ερωταποκρίσεων. Okay. English. Δεν υπάρχει διερμηνία στα αγγλικά για κάποιο λόγο. Αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα.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 κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Καλά. Continue in English? You can try continuing in English and we'll see if the French is there. Okay. Θα συνεχίσω λοιπόν στα αγγλικά. Well, then let's do it in English and uh, it, it is... Ας συνεχίσουμε στα αγγλικά για να δούμε αν θα υπάρχει τώρα τεχνικό πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε την πιο σημαντική φυσική καταστροφή μέχρι τώρα στο Πακιστάν. Πάνω από 20 εκατομμύρια άτομα έχουν πληγεί από την κρίση. Η κυρία Γεωργίεβα, επίτροπος υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια, πήγε στο Πακιστάν την περασμένη εβδομάδα και θα μας ε, πει ε, συνοπτικά αυτά τα οποία είδε επί τόπου. Σας δίνω κατευθείαν το λόγο και συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα συνεχίσω κι εγώ στα αγγλικά, αφού υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην αρχή με τα γαλλικά. Ήθελα μάλιστα να πω στην Επιτροπή ότι κάνω μαθήματα γαλλικών και έχω προοδεύσει αρκετά στα γαλλικά μου, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο μεγάλες οι προόδοι ώστε να εκτεθώ στα γαλλικά ενώπιόν σας σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την Επιτροπή για αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Είναι τεράστια η καταστροφή. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ εν συντομία με τον πρέσβη του Πακιστάν και ξέρω ότι για το λαό του Πακιστάν η σημερινή μας συνεδρίαση είναι ένα σύμβολο της υποστήριξης ε, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιο συγκεκριμένα. Και είναι ε, επίσης ένα σύμβολο της υποστήριξης ε, για αυτούς ε, που δουλεύουν επιτόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα ο στόχος μου είναι να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου από το ταξίδι μου στο Πακιστάν και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα στις προσπάθειές μας. Ακόμη, θέλουμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα από αυτή την ε, πρόσφατη καταστροφή και στρέφομαι σε εσά, τα μέλη της Επιτροπής, για να μου πείτε τις συμβουλές που εσείς έχετε να μας δώσετε. Οι εντυπώσεις μου από το Πακιστάν καταρχήν. Θα ήθελα ε, να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας το σύντομο ιστορικό των πλημμυρών που ξεκίνησαν τέλος Ιουλίου και ήταν ιδιαίτερα σφοδρές. Από τις 26-27 Ιουλίου μέχρι τις 29 Ιουλίου ε, έγιναν οι πρώτες έντονες πλημμύρες ε, και σκοτώθηκαν 1.200 άτομα στο βορρά, εκεί δηλαδή όπου ξεκίνησε αυτή η φυσική καταστροφή. Οι υπηρεσίε της Γενικής μας Διεύθυνσης ε, της ΕΚΟ ε, χορήγησε 30 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Ιουλίου, λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά τα χρήματα ε, ήταν για το Χάιμπερ και στις ομοσπονδιακά διαχειριζόμενες περιοχές του Πακιστάν και χορηγήθηκαν τελικά για την ανακούφιση των πλημμυρών. Έκτοτε οι πλημμύρες επεκτάθηκαν προς τον Νότο μέχρι και τη θάλασσα. Και όπως θα έχετε δει και από την τηλεόραση, είναι τεράστιες οι επιπτώσεις για τη ζωή εκατομμυρίων ατόμων. 17,6 εκατομμύρια άτομα έχουν πληγεί σύμφωνα με τις αρχές του Πακιστάν, εκ των οποίων πάνω από 8 εκατομμύρια χρειάζονται άμεση βοήθεια. 1,2 εκατομμύρια οικίες έχουν είτε καταστραφεί είτε πληγεί 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκταση που έχει πλημμυρίσει. Μια έκταση μεγαλύτερη από την επιφάνεια της Αγγλίας ή ας πούμε ότι είναι πενταπλάσια της επιφάνειας του Βελγίου για να έχουμε μια εικόνα της καταστροφής. Σύμφωνα με τον Πακιστανό Υπουργό Γεωργίας, 1,42 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί και σύμφωνα με, τις διεθν... με τους διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Αναπτυξιακή Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών θεωρούν ότι οι επιπτώσεις επί της ε, γεωργικής έκτασης είναι πολύ υψηλότερες και λένε ότι έχουν πληγεί πάνω από 3,4 εκατομμύρια εκτάρια. Και το πιο δύσκολο έργο είναι το να φτάσουμε στους ανθρώπους αυτούς που είναι πλήρως αποκομμένοι από τη βοήθεια είτε διότι έχουν καταρρεύσει οι υποδομές, δεν υπάρχουν πια οδικά δίκτυα, δεν υπάρχουν γέφυρες, είτε διότι έχουν περιτριγυριστεί από το νερό των πλημμυρών. Και ο αριθμός αυτών των ατόμων είναι πάρα πολύ υψηλό. Μιλάμε πάνω, για πάνω από 800.000 άτομα στα οποία δεν έχουμε καν πρόσβαση. Αν λοιπόν συγκεντρώσετε όλα αυτά τα στοιχεία που σας έδωσα, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι οι επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πακιστανικές αρχές και οι ανθρωπιστικέ οργανώσει που επιτόπου προσπαθούν να βοηθήσουν προσπαθούν να επικεντρωθούν στι άμεσε προτεραιότητε, δηλαδή νερό, φαγητό, υγιεινή, καταφύγιο, κυρίως σκηνές, ως παροχή βοήθειας. Και είναι ηρωνικό ότι για ανθρώπους που περιβάλλονται από νερό, από την πλημμύρα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Την τελευταία εβδομάδα ήδη είδαμε ότι διαδίδονται ασθένειες που μεταδίδονται από το νερό και αν αρχίσουν να εξαπλώνονται ασθένειες θα είναι τέτοια ε, η καταστροφή που θα δημιουργηθεί πολύ δύσκολη κατάσταση για, τους, για το λαό του Πακιστάν γενικότερα. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω ήδη τα κράτη-μέλη που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Κέντρου Παρακολούθησης και Ενημέρωσης για τη συντονισμένη βοήθεια ακριβώς διότι αναγνώρισαν την ανάγκη για πόσιμο είδωρ και έδωσαν πολλές μονάδες καθαρισμού του ύδατος καθώς και δισκία καθαρισμού του ύδατος. Ξέρουμε ότι τις τελευταίες μέρες ε, λίγο υποχώρησε το νερό των πλημμυρών, στο βορρά περισσότερο από ότι στο νότο. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι σίγουρη ότι η κρίση έχει φτάσει στο χειρότερο σημείο της και αυτοί που δουλεύουν επιτόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια αναφέρουν ότι τώρα έχουν πληγεί περίπου 2 εκατομμύρια ε, και έχουν ε, λάβει βοήθεια τα 2 εκατομμύρια, ενώ το σύνολο αυτών που έχουν πληγεί είναι 8 εκατομμύρια περίπου. Επεκτείνεται η κρίση και ίσως να χειροτερέψει ακόμη η κατάσταση πριν αρχίσει να βελτιώνεται. Παρότι υποχωρεί το νερό, αν ανοίξετε τις εφημερίδες σήμερα θα δείτε ότι οι ειδήσει στο Πακιστάν αναφέρονται στο κρίκετ και όχι στις πλημμύρες. Η κύρια λοιπόν εντύπωσή μου από την, από την επίσκεψή μου στο Πακιστάν είναι ότι αυτό που δυσκολεύει τόσο πολύ την κατάσταση είναι ότι έχουμε ταυτόχρονα δύο καταστροφές. Στο βορρά αντιμετωπίζουμε και τις ε, διενέξεις που υπάρχουν και τα, ε, τους εσωτερικά εκτοπισμένους ε, από το Αφγανιστάν, οι οποίοι έχουν πληγεί και από τις πλημμύρες, επομένως έχουν πληγεί δύο φορές, και στο νότο βλέπουμε ότι έχουν καταστραφεί σπίτια έχουν καταστροφεί ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και οι επιπτώσεις στη γεωργία που του χρόνου, την επόμενη περίοδο εμπορίας, ενδέχεται να τους επηρεάσουν ακόμη χειρότερα. Δηλαδή πλήττονται σήμερα από τις πλημμύρες και τους επόμενους μήνες μπορεί να πληγούν από επιστημιστική κρίση. Επισκέφτηκα το βορρά του Πακιστάν, όπου έχουμε δώσει βοήθεια σε θύματα σειράξεων και σε εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, πήγα σε ένα χωριό πλήρως κατεστραμμένο στην περιοχή Νοσέρα, όπου το μεγαλύτερο, πλήθος, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Μίλησα με κάποιον ο οποίος είχε έρθει σε αυτό το χωριό στο Αζαχέλ προσπαθώντας να ξαναστήσει τη ζωή του, αλλά τον, τον Ιούλιο καταστράφηκε το σπίτι του, όπως και το υπόλοιπο χωριό, και όταν υποχώρησε το νερό, μόνο λάσπη είχε μείνει πίσω. Λάσπη και σπασμένα ξύλα από τα σπίτια τους. Όπως λοιπόν και άλλα θύματα στο βορρά, η οικογένειά του είχε πληγεί δύο φορές και από την ε, σύραξη επιτόπου ε, και στο Αφγανιστάν και από τις πλημμύρες ε, τώρα τον Ιούλιο. Και όταν έμαθε πια ήμουν, μου μίλησε σε πολύ καλά αγγλικά και μου έκανε μία άμεση ερώτηση. Τι θα κάνει η Ευρώπη για να μας βοηθήσει. Για το δικό του το χωριό είχα μια απάντηση. γιατί προσπαθούμε να δώσουμε χρήματα ούτω ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι, να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους και να ξαναδημιουργήσουν τη ζωή τους. Άρα για το δικό του το χωριό μπορούσα να του πω τι κάνουμε. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων ενώ έχουν πληγεί 8 εκατομμύρια από τις ε, πλημμύρες και για πάρα πολλά άλλα χωριά χρειάζεται βοήθεια. Χαίρομαι που υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που ασχολούνται με την, με την ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου, προσπαθούμε για όλα αυτά τα χωριά να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Και όταν μιλάμε για πρόσβαση σε όλα τα θύματα των πλημμυρών, δεν είναι μόνο ε, θέμα φυσικής προσέγγισης, αλλά υπάρχουν και θέματα ασφάλειας και πολλές φορές ε, έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, δηλαδή ότι ε, πρέπει να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση ε, όσον αφορά την οδική πρόσβαση, αλλά πρέπει να υποστηρίξουμε και τα θέματα ασφάλειας για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα θύματα. Να πούμε λοιπόν τώρα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση ΑΕΚΟ για ό,τι έχουν κάνει και εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που μέρα και νύχτα δουλεύουν επί τόπου και τους είδα εκεί στο Πακιστάν να αγωνίζονται. Εκτός από τα 30 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν στις 31 Ιουλίου ως βοήθεια για το Πακιστάν, έχουμε και μια νέα απόφαση για 40 εκατομμύρια ανθρωπιστικής βοήθειας, πράγμα που φτάνει την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα 70 εκατομμύρια. Έχουμε κινητοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και στις 6 Αυγούστου στείλαμε μια πλήρη ομάδα και την ομάδα που στέλνουμε, η ομάδα που στέλνουμε ε, είναι ομάδα που συντονίζει την ευρωπαϊκή βοήθεια όλων των κρατών μελών. Από Σουηδία, Γερμανία ε, ε, στάλησαν ε, μονάδες καθαρισμού του ύδατος, από την Ιταλία και την Ουγγαρία φάρμακα, τρόφιμα από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Σλοβακία και Γαλλία άλλο υλικό όπως σκηνές παραδείγματος χάρη. Και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, γιατί με προθεσμία μιας ημέρας ε, έδωσε την έγκρισή του ε, για την απόφαση ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη βοήθειά μας από 10 σε 40 εκατομμύρια. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για τους ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθεια άμεσα. Αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, επισήμως θα είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα. Και έχοντας δει αυτά τα οποία συμβαίνουν επί τόπου στο Πακιστάν, τα 70 εκατομμύρια έχουν ε, ήδη αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεων, ε, έχουν συμβασιοποιηθεί και δεν θα είναι και αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε γρήγορα, διότι έχουμε επιτόπου εμπειρογνώμονες και αυτοί οι εμπειρογνώμονες ήδη είχαν συνεργαστεί στενά με τις πακιστανικές αρχές μου έκανε εντύπωση ο στρατηγό Αναποστατή Αναντίμ, επικεφαλής τη Εθνική αρχή διαχείριση ε, της κρίσης στο Πακιστάν και δούλευε με το επιτελείο του με περίπου 23 άτομα για να συντονίσει όλες τις περιφερειακές αρχές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εκείνος και άλλοι επικεφαλεί των αρχών ε, παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι στο Πακιστάν και ε, χωρίς την εξωτερική βοήθεια, τη βοήθεια τη δική μα δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με μια τέτοια καταστροφή. Τα κράτη-μέλη ανταποκρίθηκαν ε, πολύ γρήγορα στην έκκληση να εντείνουν τη βοήθειά τους και σήμερα οι δεσμεύσει ε, των κρατών μελών φτάνουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί λοιπόν με την Επιτροπή έχουμε δώσει 230 εκατομμύρια ευρώ, 320 εκατομμύρια δολάρια δηλαδή είχαν ζητήσει αρχικά τα Ενωμένα Έθνη 460 εκατομμύρια δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε ανταποκρίνεται νεόδωρα και μάλιστα τα καταφέραμε και πάρα πολύ γρήγορα με σημαντική βοήθεια. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει. είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια με μέτρα ανάκαμψης, πρώης ανάκαμψης. Και εδώ θα πρέπει να ασχοληθούμε με μέτρα που αφορούν τη γεωργία, γιατί καθώς υποχωρεί το νερό των πλημμυρών στο βορρά, για να μην χάσουμε αυτή την εποχή σποράς, θα χρειαστούν ε, ταχύτατα και σπόροι προσφορά και γεωργικά εργαλεία για τους αγρότες και στο βορρά αλλά και στο νότο για να μπορούν να φυτέψουν τη νέα σοδιά. Και είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθούν οι κρίσιμες συνδέσεις στο δικό δίκτυο με γέφυρες και δρόμους και για να μπορούμε να φτάσουμε στα θύματα, αλλά και να μπορούν να συνδεθούν οι αγρότες με την αγορά. Γιατί όταν ταξιδεύει κανείς στο Πακιστάν είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στις περιοχές που έχουν πληγεί από την πλημμύρα και στις περιοχές ακριβώς δίπλα σε αυτές. Ακόμη και 100 μέτρα μπορεί να να δίνουν τεράστια διαφορά τελικά. Δηλαδή υπάρχουν χωριά και πόλεις που έχουν πληγεί και δίπλα τους υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν πληγή. Είναι λοιπόν τεράστια σημασία του να υπάρξει υποδομή, να αποκατασταθούν οι υποδομές που έχουν καταστραφεί για να μπορέσει να ορθοποδήσει και πάλι η χώρα. Μακροπρόθεσμα, θα χρειαστεί ε, να αποκατασταθούν οι υποδομές και να αποκατασταθεί η χώρα και κοινωνικο-οικονομικά. Η Διεθνής Τράπεζα, ε, η Υπηρεσία Ανάπτυξη των Ηνωμένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζουν την αξιολόγηση αναγκών που θα χρειαστεί 4 έως 6 εβδομάδες ακόμη μέχρι να ολοκληρωθεί. σε αυτή την μακροπρόθεσμη ανάκαμψη θέλω να τονίσω δύο σημεία. Καταρχήν το πόσο κρίσιμη είναι η συνεργασία και ο συντονισμός. Είναι κέρια σημασία και απαιτείται συλλογική προσπάθεια η οποία πρέπει να καταβληθεί με συντονισμένο τρόπο. Και κάτι άλλο πιο σημαντικό ακόμη κατά τη γνώμη μου. Το Πακιστάν είναι από τις πλέον ευπαθείς ως προς κλιματικές αλλαγές ε, χώρες ε, και έχει ταξινομηθεί βάσει κάποιων δικτών ε, ως πλέον ευπαθείς πάντα ως προς τις κλιματικές αλλαγές. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε την, α, τις δράσεις ανακούφισης και αποκατάστασης με τρόπο ώστε να είναι προετοιμασμένο το κράτος αυτό για την επόμενη καταστροφή. Δεν, ε, κανείς δεν αποδεικνύει ότι οφείλονται σε κλιματικές αλλαγές αυτές οι πλημμύρες, αλλά οι επιστήμονες κατηγορηματικά ισχυρίζονται ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών ε, φαινομένων οφείλεται σε κάθε περίπτωση στις κλιματικές αλλαγές. Ε, χρειάζεται αναδάσωση, αποκατάσταση των ανθρώπων σας είπα ότι έβλεπα ανθρώπους που ζουν σε σπίτια κατεστραμμένα που όμως φαίνεται ότι ούτως ή άλλως ήταν ακατάλληλα εξ αρχής. Όλα αυτά τα μέτρα που αναλαμβάνουμε θα μας αποδώσουν ηγετικό ρόλο και έτσι επιβεβαιώνεται η επεποίθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όχι μόνο θα μειώσουμε τις εκπομπές για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές αλλά και θα επιδιώξουμε ενισχυμένη δράση σε, ε, στις πιο ευπαθείς χώρες όπως το Πακιστάν. Ω προ ε, την ε, αρρωγή προς το Πακιστάν, ε, θα ήθελα να σα πω ότι εξεπλάγει θετικά από τι επαφέ που είχαμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν σχετικά με την λογοδοσία για τα κονδύλια που καταβάλουμε στο Πακιστάν. Προάγουν την διαφάνεια για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων και συστάθηκε και η Ειδική Επιτροπή που θα επιβλέπει την εξωτερική βοήθεια και με ρώτησαν μάλιστα ε, αν έχω κάποιες ε, ιδέες ε, για να αναβαθμιστεί η διαδικασία ως προς τη διαφάνεια δηλαδή και τη λογοδοσία για τα κονδύλια που προέρχονται από το εξωτερικό. Ε, φυσικά πρέπει να έχουμε ε, εμπιστοσύνη στο Πακιστάν. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι η μόνη πληγή από φυσικές καταστροφές χώρε, γιατί ως επικεφαλής υπηρεσίας μου ε, σας λέω ότι ανησυχώ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η περίοδος των τυφώνων και φοβούμε και για άλλες χώρες και ο τελευταίος χρόνος ε, έχει δει αλλεπάλληλες ε, καταστροφές σε διάφορες χώρες. Πάντως ε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτω ώστε το έπακρο να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Τον ερχόμενο μήνα θα σας υποβάλουμε εκ νέου αναφορά Ε, για να σας μιλήσουμε για το μέγεθος καταστροφής και για τη χρήση των κονδυλίων. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ποια είναι τα διδάγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. In our work we need to put much... Φυσικά ε, θα πρέπει να ε, επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην προετοιμασία για τις ε, φυσικές καταστροφές. Μόνο αν είμαστε ε, καλύτερα προετοιμασμένοι θα ε, χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικότητα τον προϋπολογισμό που έχουμε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη σας μίλησα για την κέρια σημασία του να αυξήσουμε την προετοιμασία των ευπαθών χωρών για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ε, την τελευταία δεκαετία τι διαπιστώσαμε ότι στα 9 από τα 10 χρόνια δεν είχαμε επαρκή κονδύλια γιατί είχαμε υπεράριθμες καταστροφές σε σχέση με τον προπολογισμό μας. Οπότε ε, Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ε, διαπιστώνουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Το δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε και που ε, καθορίζει δηλαδή τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να συζητηθεί. Επίσης, με την ε, Βαρόνη Άστον, με τον κύριο Πίμπαλξ και άλλους ε, συναρμοδίους επιτρόπους ε, συζητούμε το θέμα. Η ύπατη εκπρόσωπος, η Άστον και η υποφαινόμενη ήρθε σε στενή επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών Βανάκυρεν από τη Βελγική Προεδρία που μίλησε στις 9 Αυγούστου ε, σχετικά με τις ε, θετικές, ε, τη θετική αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις κρίσης. Παρά τις προσπάθειες όμως που κάνουμε, βλέπουμε επικριτικά δημοσιεύματα στον τύπο και το αναφέρει πόσο σημαντική είναι και η επικοινωνιακή μας πολιτική. Δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα ανταπόκριση Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρούμε με συντονισμένο τρόπο και να χρησιμοποιούμε ε, συλλογικά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Ε, Κλείνοντα. Θα έλεγα ναι, πως ναι, είναι τραγική αυτή η φυσική καταστροφή, αλλά είναι και ευκαιρία για να καταδείξουμε αλληλεγγύη, να καταδείξουμε ότι έχουμε κοινέ αξίες που μας ενώνουν η αλληλεγγύη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά μεταφράζεται σε δράσεις και μέσα από αυτές τις δράσεις θα φέρουμε την αλλαγή στην καθημερινή ζωή αυτών των ε, πλημμυροπαθών. Θα εργαστούμε άκνα, ούτως ώστε να ε, διατηρήσουμε ε, και να ε, παράσχουμε με συντονισμένο τρόπο τη βοήθεια από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσουμε τους, τον πληθυσμό του Πακιστάν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε και τους εξής, τα εξής πρόσωπα, τον κύριο ε, Αντουάν από την ΟΚΑ Τέρμαν Κάτι, UNICEF, Σάιμον Μισήρ, ε, διεθνή Συνομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, Φρανσουά Μπέλα, ε, διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και Κάτριν Σίκ από το Voice. Θα ήθελα και εκείνοι να παρέμβουν κατά, το, κατά τη λήξη της συζήτησης. Έχουμε δέκα μέλη που ζήτησαν το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να είστε ιδιαίτερα σύντομοι, δηλαδή να μιλήσετε για δύο λεπτά έτσι ώστε να μπορέσετε όλοι να λάβετε το λόγο πριν δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να συνοψίσει. Ο κύριος Μίτσελ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την έγκαιρη απάντησή της και για τη δράση της. Χαίρομαι για τη δράση που αναλήφθη και θα ήθελα να συνεχίσει αυτή τη δράση. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε από πού θα αρχίσουμε. Αν δεν ανταποκριθούμε θα πεθάνουν πολλοί κατά εκατοντάδες. Είχαμε ε, μεγάλα προβλήματα στη, στο βορρά της περιοχής, της χώρας και ε, βεβαίως ε, γνωρίσαμε και εκτός από τις ε, πλημμύρες και σεισμούς και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε και άλλες ε, εύπορες χώρες της περιοχής να συνεισφέρουν. Πολλοί φαίνεται ότι μένουν πίσω. Θα πρέπει να πιέσουμε όλες τις χώρες να αναλάβουν δεσμεύσεις. Και νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το θέμα στο προσκήνιο και όταν φύγει από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Το θέμα που έθιξε η Επίτροπος για ολοκλήρωση και συντονισμό, αυτό το θέμα είναι ουσιώδες. Θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων μας και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να εστιάσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στην προστασία των πληγέντων, αλλά και στις ευάλωτες ομάδες και σε αυτούς που διατρέχουν μεγάλους κινδύνους. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι θέμα μόνο ε, βοήθειας, θα πρέπει να βοηθήσουμε και προς την ανάκαμψη και να βοηθήσουμε τους πληγέντες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, θα δώσω το καλό παράδειγμα επανήλθαμε μετά το καλοκαίρι, γιατί αυτή είναι, αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας και θα πρέπει να το θέσουμε στο επίκεντρο των σκέψεών μας. Ελπίζω να ανταποκριθούμε στις ε, δεσμεύσεις και θα πιέσουμε και άλλους να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Αυτό θα είναι ένα απόσπαθο τμήμα της στρατηγικής μας. Ο κύριος Γκερέιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί καταβάλατε προσπάθεια προσωπικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει καταρχήν να τονίσω ότι με εξέπληξε η αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών εναντί αυτού του δράματος, ιδιαίτερα αν την συγκρίνουμε με την αντίδραση, την άμεση αντίδραση στην περίπτωση της ΑΙΤΙΣ. Επειδή ανέκυψαν ε, και οι καλοκαιρινές διακοπές και επειδή αυτή η χώρα είναι πιο μακρινή και με την οποία γνωρίζουμε θρησκευτικές διαφοροποιήσεις δεν σημαίνει ότι την αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δράμα των ανθρώπων και θα πρέπει να το κάνουμε σε επίπεδο αρχών όπως κάνουμε σε κάθε περίπτωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει να είναι ουδέτερη και αμερόληπτη η βοήθειά μας, ανεξάρτητη και να συνάδει με τις ανάγκες της περιοχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν ίσχυσε. Θα πρέπει να είναι ορατή η βοήθειά μας, διότι αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν άλλοι. Και τα προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται θα έχουν αντίκτυπο σε εμάς τους ίδιους. Θα ήταν παράλογο να αγνοήσουμε το θέμα πολιτικής σταθερότητας που αντιμετωπίζει το Πακιστάν και την ε, γεωστρατηγική του σημασία ως προς τις ε, δημοκρατικές αξίες ανά τον κόσμο. Γι' αυτό νομίζω ότι με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να υπάρχει μια ε, δημοκρατική ορατότητα μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ. Η παρούσα καταστροφή θα πρέπει να οδηγήσει σε μια δίχρονη αντίδρασή μας. Καταρχήν θα πρέπει να ανταποκριθούμε στα άμεσα, να προβάλλουμε μια άμεση βοήθεια και η Επίτροπος ανταποκρίθηκε στην εργασία της. Σε μια ανακοίνωση τύπου με την κυρία Ζολή αυτό ακριβώς ε, τόνισα, δηλαδή ε, ανταποκριθήκατε μέσα στα πλαίσια των χρηματοδοτικών ορίων. Μπορούμε να διευρύνουμε αυτόν τον ορίζοντα αν έχουμε καλύτερο συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την παρέμβαση. Καταρχήν θα ήθελα να δείξω και το εξή. Θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις δεσμεύσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε όλες τις πρόδειλες ανάγκες του πακιστανικού λαού μέσα στα πλαίσια της ανάκαμψης. αν και άμεσα δεν μπορούμε να έχουμε άμεση χρηματοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να εγγραφούν νέα κονδύλια ή να ανοιχτούν νέες δυνατότητες, να ανοιχτούν νέες δυνατότητες. Κατά δεύτερον, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγκη. Ζούμε σε μια κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου για πολλούς. Αυτή η καταστροφή θα πρέπει να μας καταδείξει ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Έχουμε την έκθεση Μπαρνιέ και αρκεί να τη θέσουμε σε εφαρμογή. Δεν έχουμε κανένα ελαφρυντικό για να μην ανταποκριθούμε έναντι αυτής της καταστροφής ως προς ε, θέμα καθαρά ορατότητας. Νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Δεν το προσάπτω σε ε, εσάς αυτό. Δεν μιλάμε για ε, προμελετημένη γενεοδορία. Αλλά νομίζω ότι οι πρωταρχικοί δωρητές δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί τη στιγμή που ζούμε σε μια κατάσταση άμεσης καταστροφής. Θα ήθελα να γίνει μια σύσκεψη και έπρεπε ήδη να έχει γίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών για να καταδείξουμε στους Πακιστανούς ότι πρέπει να ανταποκριθούμε. Λυπάμαι, λέει η πρόεδρος, δεν μπορείτε να συνεχίσετε, υπάρχει περιορισμός ο χρόνο. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση ad hoc για τη διερμηνία και ελπίζουμε να την έχουμε για την διερμηνία προς τα αγγλικά. Έτσι θα δοκιμάσω και τα γαλλικά, μου λέει η Επίτροπος. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ανταποκριθώ ως προς την διαθεσιμότητα κονδυλίων, να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε ως προς την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Στην Ολλανδία Έχουμε προγράμματα στην τηλεόραση για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και, το δύο, και μαζέψαμε 16 εκατομμύρια. Το 2005 σε ε, ένα σεισμό στο Πακιστάν είχαν συλλεγεί 85 εκατομμύρια. Επίσης για την IT 111 εκατομμύρια συλλέξαμε πέρσι. Αυτά ήταν τα ποσά. Άρα πιστεύω ότι η Ολλανδία μάζεψε πολύ, ε, μάλλον δεν ανταποκρίθηκε στον ίδιο βαθμό, γιατί μαζέψαμε πολύ λιγότερα χρήματα ε, φέτος για την παρούσα κρίση. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εγγραφούν νέα κονδύλια, αυτό είναι απόλυτα σαφές. Άκουσα την Επίτροπο, άκουσα την παρέμβαση της Επιτρόπου, η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχουν πλέον κονδύλια, δεν έχει τελειώσει και η περίοδος των μουσώνων πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στην παρούσα κρίση. Πώς, ε, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που επιβάλλεται. Θα ήθελα μία εντελεχέστερη ανάλυση από την δική σας πλευρά επί του θέματος. Δεν σημαίνει ότι δεν ε, εμπιστευόμαστε τις πακιστανικές αρχές ως προς το σκέλος της ανοικοδόμησης. Αυτό ήδη προαναφέρθηκε. Θα ήθελα όμως να ακούσω το εξής. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάκαμψης μέσα στα πλαίσια εκδημοκρατισμού της χώρας. Μιας χώρας που αντιμετωπίζει μεγάλα και θρησκευτικά προβλήματα και πολιτικά και σύραξης με το Αφγανιστάν. Υπάρχουν διάφορες βομβιστικές ενέργειες Υπάρχει το θέμα, το πρόγραμμα του αλφαβητισμού και των σχολείων. Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στο θέμα αυτό. Ο κύριος Λαμπέρ, η κυρία Λαμπέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, λαμβάνω το λόγο ω Πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Νοτιοανατολική Ασία και συμπεριλαμβάνεται και το Πακιστάν στι χώρε αυτέ χαιρετίζουμε την ανταπόκριση της Επιτροπής στην καταστροφή στο Πακιστάν και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας ε, ε, προς το λαό του Πακιστάν μέσω του πρέσβη που είναι παρόν. Ε, έχω ένα ερώτημα, όχι τόσο για την άμεση αρρωγή που προσφέρεται, αλλά περισσότερο όσον αφορά την αναδιάρθρωση της χώρας. Συμφωνώ πολύ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα κατά τη φάση ανασυγκρότηση. Αλλά θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει το ζήτημα του διεθνούς χρέους του Πακιστάν. Πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι η αποπληρωμή αυτού του χρέους θα, είναι, θα αφορά μεγαλύτερο ποσό από τα ποσά τα οποία φτάνουν στο Πακιστάν ως βοήθεια και γι' αυτό θα ήθελα ε, να εξετάσει η Επιτροπή το αν είναι δυνατόν να υπάρξει είτε μερική ακύρωση αυτού του χρέους είτε κάποιο, κάποια στάση του χρέους ε, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Γιατί θα φτάνουν τα χρήματα τη δική μας βοήθειας προς το Πακιστάν, αλλά δεν θα έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, διότι η κυβέρνηση του Πακιστάν θα πρέπει να αποπληρώνει το παλαιό τη χρέος. Και χαιρετίζω τα μηνύματα τα οποία μας μεταφέρατε σήμερα για την πρωτοβουλία διαφάνειας, διότι σίγουρα πολλοί από τους δωρητές έχουν τέτοιες ανησυχίες που αφορούν τη διαφάνεια. Και συμφωνώ επίσης ότι πρέπει και άλλες χώρες να ενθαρρυνθούν, όχι μόνο οι χώρες ε, της περιφέρειας, και άλλες χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να δώσουν βοήθεια και κυρίως ε, χρήματα ε, και θα αποφασίσει από εκεί πέρα το Πακιστάν το πώς θα δαπανηθεί αυτή η βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Κόβατσεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για όσα μας είπατε για την κατάσταση στο Πακιστάν και για τις δράσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό και για τα δύο θεσμικά όργανα και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και να διευκολύνουμε η ΜΕΝ το έργο των ΔΕ ε, για κρίσεις όπως αυτή η κρίση στο Πακιστάν. Είναι μια ανθρωπιστική, βοήθεια, ε, μια ανθρωπιστική καταστροφή που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και για το Πακιστάν είναι τεράστια αυτή η καταστροφή και αν το δούμε σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως η δική μου χώρα είναι τεράστια η επιφάνεια που πλήττεται από τις ε, πλημμύρες και επομένως χρειάζεται άμεση βοήθεια και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεταξύ των πρώτων που βοηθούν σε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή. Ευχαριστούμε την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα και το προσωπικό της Επιτροπής για την βοήθεια την οποία φροντίσατε να δώσει η Επιτροπή. Δουλεύουμε σε αλληλεγγύη προ το λαό του Πακιστάν. Η Επιτροπή, όπω είπατε, ήταν η πρώτη που αντέδρασε υπέρ αυτή τη καταστροφή και παρότρινε τα κράτη-μέλη ώστε συνολικά να συγκεντρωθούν ε, πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια. Α είμαστε όμω ε, ειλικρινεί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση, ιδιαίτερα στο βορρά τη χώρα και γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ο πληθυσμό του Πακιστάν και οι πρόσφυγε από το Αφγανιστάν που έχουν πληγεί δύο φορέ, όπω είπατε, και πλήττονται και από τι πλημμύρε και από πλευρά ασφαλεία. Πλήττονται διότι από του εξτρεμιστέ συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο και ε, όλοι φοβούνται ότι υπάρχει ο κίνδυνο αποσταθεροποίηση λόγω των εξτρεμιστών και για το Πακιστάν και για το Αφγανιστάν, τη γειτονική χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ξέρετε ότι εμεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρέχουμε τη βοήθειά μα. Ευχαριστώ. Merci Θα ευχαριστούμε. Ο κύριο Βότσον ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αρχίζουμε, συζητούμε για τα πρώιμα στάδια της ανακούφισης δεδομένη στις βαρύτας της ε, ε, κατάστασης. Βέβαια αληθεύει ότι υποχωρούν τα νερά, αλλά οι μετεωρολογικές ε, προβλέψεις σαφώς δείχνουν ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτό για 10 με 12 μέρες. Στην περιοχή ΣΥΝΤ βέβαια φαίνεται ότι δεν θα υπερχειλιστεί ο ποταμός και πάλι. Το Πακιστάν και η Ινδία εδώ και χρόνια πλήττονται από σοβαρές πλημμύρες, ε, αλλά εδώ μιλάμε για το 10% του πληθυσμού του Πακιστάν που αυτή τη φορά επλήγει Υπάρχουν ε, σημαντικές ε, ε, ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν λόγω των πλημμύρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις κοινέ προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων και μονομένες προσπάθειες και στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακούφιση του Πακιστάν. Αλλά πρέπει με ταχύτερο τρόπο να διαθέτουμε τα διαθέσιμα κονδύλια και δεδομένων των συνθήκων θα πρέπει να ε, λειτουργήσουμε με σοβαρότητα, με συντονισμένο τρόπο, δεδομένου και των κλιματικών αλλαγών. Ε, εσείς μιλήσατε για τις αλλεπάλες φυσικές καταστροφές την τελευταία δεκαετία. Ε, ε, λοιπόν, θα επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω η κατάσταση. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, διότι δυστυχώς θα γίνουμε μάρτυρες πολύ μεγαλύτερης ανθρώπινης δυστυχίας στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρύμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να καλωσορίσω την αρχική σας παρέμβαση. Ε, σας ευχαριστούμε που ε, πήγατε επί τόπου στο Πακιστάν γιατί έτσι ε, ε, μεταφέρατε ένα σαφές μήνυμα στον επιτόπιο πληθυσμό. Πρώτη ημέρα συνεδριάζουμε σήμερα και ε, φαίνεται ότι είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας το θέμα του Πακιστάν και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα στηρίξουμε το Πακιστάν για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την μείζουνα κρίση σχετικά με την, ε, την ε, επιχείρηση διάσωσης ε, που σχεδιάζουμε, αναφερθήκατε σε κάποια επιμέρους σημεία, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διτή προσέγγιση. Πρώτον, να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε στον τομέα της ανακούφισης και της ανοικοδόμησης, αλλά να έχουμε κατά νου ότι δεν θα κρατήσει η κατάσταση, δεν θα παραμείνει έτσι η κατάσταση μόνο για τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, για μήνες και για χρόνια θα πρέπει να πρωταγωνιστεί το Πακιστάν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε το Πακιστάν για την ανοικοδόμηση, για την οικοδόμηση νέων υποδομών, ε, για να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά μελλοντικέ καταστροφέ. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι πρέπει να κάνουμε, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τον πληθυσμό του Πακιστάν ε, για να βοηθήσει και ε, ο πληθυσμό του Πακιστάν την ίδια τη χώρα να ορθοποδήσει στη συνέχεια. Ε, και το Πακιστάν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές, στις αγορές συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να υπάρχουν αυξημένες εμπορικές ροές και να επικουρηθεί στις προσπάθειες που κάνει. Το 2005 μην ξεχνάτε ότι είχε ψηφιστεί ένα σχετικό ψήφισμα όπου λέγαμε ότι υποστηρίζουμε το άνοιγμα, το μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών προς το Πακιστάν. Ε, είχε αντιδράσει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να απευθύνω αυτή την να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα του Κοινοβουλίου προς τους συναδέλφους σας, τους λοιπούς ε, επιτρόπους. Ευχαριστούμε κύριε Καρύμ, ο κύριος Ελμαμπρόκ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. από τότε που αρχίσατε τις ε, αρμοδιότητες σας ως Επίτροπος έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να τα βγάλετε πέρα γιατί αντιμετωπίσατε πολλές ε, καταστροφές. Στο Πακιστάν έχουμε πολλές ε, ε, καταστροφές. Έχουμε το, το πρόβλημα των Ταλιμπάν και των προβλημάτων ασφαλείας στην περιοχή. Έχουμε το πρόβλημα του ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πείνα και την επιστημιστική βοήθεια που πρέπει να χορηγηθεί ε, και πρέπει ε, κατά τρίτον ε, να φροντίσουμε ώστε να είμαστε αρκετά γρήγοροι ώστε να φτάσει η ανθρωπιστική μας βοήθεια επιτόπου πριν να περάσει από τους Ταλιμπάν. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε το πώς ε, θα διεξάγεται η όλη διαδικασία. Και είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ε, τις διαθρώσεις που απαιτούνται ε, και πολύ γρήγορα να φτάνουμε με αεροπλάνα ή με ελικόπτερα, ούτως ώστε να διασφαλίζουμε τη χορήγηση των πόρων. και ο κύριος Σαρκοζή είπε ότι χρειάζεται να χωρηθεί ε, βοήθεια επιγόντως και θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να συντονιστεί με ε, τους εθνικούς εκπροσώπους ώστε η αλυσίδα της εφοδιαστικής ε, να προχωρήσει και να φτάσουμε πιο γρήγορα ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Νομίζω αρκούν αυτά, διότι δεν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, Επίτροπο για την παρουσία της και για όσα μας είπε. Εμείς στην ουσία δεν ήμασταν παρατηρητές αυτής της μεγάλης καταστροφής και δράσαμε με μεγάλη βραδύτητα. Βεβαίως συμμερίζομαι την ανάγκη βελτίωσης της δυνατότητας παρέμβασής μας σε περίπτωσης καταστροφής και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές βοήθειας προς το Πακιστάν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Θα ήθελα όμως να μας απασχολήσει και κάτι άλλο ως προς την κατάσταση αυτή, διότι βρίσκεται εκτός ε, κάθε συζήτησης που γίνεται για τις κλιματικές αλλαγές. Ίσως θα έπρεπε να ενταχθεί όμως και εδώ, διότι θα πρέπει να προσαρμαστούμε στις ε, κλιματικές αλλαγές. Και αυτό το λέω για όσους μεταβούν στο Κανκούν ή στο Johannesburg του χρόνου. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να φτάσουμε σε ένα σύστημα ελέγχου των εκπομπών έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε πόρους για να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές μελλοντικά και αυτό με προληπτικά μέτρα για κάθε τετραγωνικό. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν. Διαφορετικά αυτές οι καταστροφές θα επιδεινώνονται ολαιοένα και περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η αναφορά σας. Ε, δύο σύντομες ερωτήσεις. Ε, η Ινδία, η Κίνα, η ΙΠΑ, πόση βοήθεια δίνουν στο Πακιστάν, μήπως ε, τυχαίνει να το γνωρίζετε, θα μας ενδιαφέρει να το μάθουμε. Και πριν από το θέρος, η Επιτροπή μας έστειλε αποστολή στην IT για να παρατηρήσει τις τελευταίες εξελίξεις και κάναν μια τρομακτική αναφορά ότι δηλαδή με το που φεύγουν οι κάμερες ε, βγάζουν, ε, αποσύρουν το πυροβολικό, το βαρύ πυροβολικό είπα και κατά 80% επικρατεί το χάος. Ε, και γι' αυτό σας ρωτάω ποιος θα ασχοληθεί με την μακροπρόθεσμη βοήθεια του Πακιστάν για να μεριμνήσουμε ώστε να μην τους εγκαταλείψουν όλοι με το που θα αποχωρήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κύριο Σαρσένης τώρα. Thank you very much, Madam Chairman. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Επίτροπε. Και σας συγχαίρω για την άμεση και ιδιαίτερα υπεύθυνη ανταπόκρισή σας στην κρίση. Επίσης σας συγχαίρω διότι προσπαθείτε να λάβετε υπόψη σας τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το κλίμα και την αναδάσωση. Μιλήσατε για τους πόρους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης και παράλληλα, εκτός από τη χορήγηση πόρων, συμφωνώ και με την ιδέα της συναδέλφου της κυρίας Λάμπερτ ότι κάτι πρέπει να γίνει και σχετικά με το χρέος του Πακιστάν. είτε να διαγραφεί μέρος του χρέους, είτε να γίνει κάποια στάση πληρωμών. Ε, αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα ε, και αναμένουμε ότι η κατάσταση του κλίματος ε, θα επιδεινωθεί περισσότερο. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε την απάντηση της Επιτροπής για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήδη λαμβάνονται μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση και όπως είπε ήδη ο κύριος ε, Πρόντι, αν δεν σταματήσουμε την ε, κλιματική αλλαγή δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να σταματήσει η συσσόρευση αερίων του θερμοκηπίου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα των αερίων του θερμοκηπίου που ήδη έχουν συσσωρευτεί και θα πληγούμε από αυτά τα αποτελέσματα μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ, όπως ε, και οι προηγούμενοι ομιλητές, να συγχαρώ την Επίτροπο, κυρία Γεωργίευα, για την ε, ταχεία και αποτελεσματική παρέμβασή της. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ε, παγκόσμιας συντονισμένης δράσης για αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή. Αν επιτόπου, δηλαδή στο Πακιστάν, είδατε τέτοιες ενδείξεις ε, διεθνού συντονισμού. Δυστυχώς αυτές οι τεράστιες καταστροφές θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι τελευταία καταστροφή αυτή που βλέπουμε. Το θέμα είναι αν μπορούμε ε, να οργανώσουμε σωστά κάποιο παγκόσμιο μηχανισμό ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και όταν προσπαθούμε να χορηγούμε βοήθεια να μην δημιουργείται σύγχυση επιτόπου αλλά να συντονίζονται οι προσπάθειες όλων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ε, καλό θα ήταν να μην πολιτικοποιούμε αυτή την παρέμβαση και την ανθρωπιστική βοήθειά μας προς το Πακιστάν. Οφείλουμε να χορηγήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες. Thank you, uh, Commissioner, for all what... Ε, ευχαριστώ, Επίτροπε, για ό,τι καταφέρατε στον τελευταίους, στο τελευταίο μήνα και ό,τι μας είπατε σήμερα. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για πολιτική παρέμβαση και στρατιωτική παρέμβαση, έτσι ώστε η αρρωγή να δοθεί στους πληγέντες. Ε, μιλήσατε και για εμπόδια και ο πρόεδρος Μπαρόζο στο γράμμα του προς τον κύριο Σαρκοζή το ανέφερε αυτό. Ως προς τη μακροχρόνια αρρωγή και ανοικοδόμηση το συζητήσατε με την κυβέρνηση του Πακιστάν ως προς το θέμα λογοδοσίας. Όμως πώς θα ε, γίνει η ανοικοδόμηση μέσα στα πλαίσια της ε, αποψήλωσης των δασών και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, μεγάλη οικολογική καταστροφή. Η κυρία Λάμπερτ μίλησε για το χρέος του Πακιστάν και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας πλαισίωσης, γιατί μιλάμε για μια χώρα που δαπανά μεγάλο μέρος του εθνικού προϋπολογισμού στο, για το στρατιωτικό σκέλος, για τις έναπλες δυνάμεις και για τα πυρηνικά, για τους πυρηνικούς ε, εξοπλισμούς. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να μεταβούν προς μία άλλη κατεύθυνση τα κονδύλια του προϋπολογισμού για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του λαού του Πακιστάν. Ο κύριος ε, Σβένσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τη διεξοδικότατη παρουσίαση που κάνατε για την εξαιρετικά επισφελή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πακιστάν. Ελπίζουμε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα γρήγορα. Χάρη που η ως μας είπε ότι υπάρχει μια δυνατότητα πλέον να καταδείξουμε πράκτος την αλληλεγγύη μας και εγώ θέλω να το τονίσω αυτό. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η καταστροφή είναι και μια θετική ευκαιρία δεν απαιτούνται μόνο πράγματα για μας, αλλά αποτελεί και χαρά για μας αυτή η ευκαιρία που έχουμε. Θα πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για τη συνολικότερη βοήθεια αλλά και για τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων στην αναπτυξιακή βοήθεια των κρατών μελών. Ε, βλέπουμε επίσης τις εικόνες ε, από το Πακιστάν, από το Αφγανίσταν, ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν τρομοκρατικές δυνάμεις, έχουμε τους Ταλιμπάν, μιλάνε για πυρηνικά όπλα. Πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε ούτως ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δείχνουν ότι με τα κονδύλια που διαθέτουμε κάνουμε κάτι θετικό για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επαρκή κονδύλια, τουλάχιστον όχι όσα θα θέλαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι τόσο μεγάλε καταστροφέ, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντεκάισερ τώρα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι σήμερα μαζί μας και που μετέβει στο Πακιστάν. Πολλοί προανέφεραν την σημασία του συντονισμού και της προβολής της δράσης και της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω να γύρω μόνο ένα ζήτημα, αυτό των γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα στο Πακιστάν. Με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον 200.000 γυναίκες ε, αναμένεται να γεννήσουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες με πιθανές, με επαπειλούμενες εγκυμοσύνες, για 30.000 γυναίκες. Είναι πελώριο αυτό το πρόβλημα και δεν έχει αντιμετωπιστεί. Οπότε ρωτώ, πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτό το θέμα, να ε, αφιερώσουμε κάποιες προσπάθειες στο συντονισμό της δράσης μας για να καλύψουμε αυτό το θέμα, για να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξει σωστή διαχείριση του ζητήματος. Εάν όχι, ε, και μην ξεχνάτε, συγγνώμη, ότι θα προβάλλουμε και την καλύτερα τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφιερώνεται στις προσπάθειες αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε κύριε Στιβέν. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα αργοπορημένη. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. μας στείλατε επιστολή όχι σε όλους τους συναδέλφους ε, με ενημερωτικά στοιχεία σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη διαθεσιμότητα που δείχνετε επί τόπου αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αυτό δεν ισχύει για όλους τους συναδέλφους σας και θέλω να το τονίσω πραγματικά. 30 ε, εκατομμύρια επιπλέον μας είπατε θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, αντιμετωπίσει την ε, αυξανόμενη σοβαρότητα της καταστροφής και συμπληρώνει αυτό τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Ε, θα πρέπει να κινητοποιηθούν επιπρόσθετα κονδύλια έκτακτης ανάγκης στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, τα μία έκτακτης παρέμβαση. Ε, η Βαρόνια Άστον μας υπέβαλε ένα έγγραφο σχετικά με τα δίδαγματα που πρέπει να αντλήσουμε από τη δράση μας στην ΑΕΤ. Ε, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στην ανακοίνωση που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου θα καταγράφει την κατάσταση σε σχέση με την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά σε έκτακτε περιστάσει και να διαχειρίζεται κρίσει. Θα υποβληθεί αυτή η ανακοίνωση το φθινόπωρο. Βέβαια, οι συνθήκε είναι λίγο διαφορετικέ στο Πακιστάν σε σχέση με την ΑΕΤ, αλλά τέλο πάντων ένα μήνα μετά ε, μπορείτε εσεί να εντοπίσετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ε, ω προ την αποτελεσματικότητα τη βοήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση, την ταχύτητα παροχή τη βοήθεια βοήθεια στο συντονισμό, την προβολή του έργου της Ένωσης. Ο μηχανισμός δε πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά ενεργοποιήθηκε. Κατά τη γνώμη σας αυτή η νέα ανθρωπιστική κρίση δεν δείχνει για ακόμη μία φορά την ανάγκη που υπάρχει να αναβαθμιστεί ο μηχανισμός. Ε, και να δημιουργηθεί ε, ο περίφημος μηχανισμός έγκαιρης ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που όπως όνεισαν και πολλοί συνάδελφοι θα οδηγήσει στην περιβόητη ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Θα δώσουμε το λόγο στους λοιπούς επισκέπτες μας για ένα λεπτό έκαστος παρακαλώ. Κατόπιν ο πρέσβης του Πακιστάν θα ε, πάρει το λόγο πριν ε, την απάντηση της Επιτρόπου σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ο κύριος Αντουάν Γεράρε, ε, για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του λαού του Πακιστάν για την άμεση αρρωγή, η οποία χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της τραγωδίας που έπληξε το Πακιστάν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Τα ενθαρρυντικά σας ε, λόγια κάνουν τη μεγάλη διαφορά υπέρ του λαού του Πακιστάν που ζει αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την άμεση αρρωγή που χορηγήσατε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκριθείτε στις πρωταρχικές ανάγκες του λαού. Ήταν μια πολύ σημαντική χειρονομία και επίσης και η σημερινή συνάντηση θα οδηγήσει σε μια υποστήριξη, γενικότερη υποστήριξη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε. Γνωρίζετε ότι ζήσαμε μια μεγάλη τραγωδία. Η εμβέλεια της καταστροφής ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και χρειαζόμαστε πολύ υψηλούς πόρους για να ανταποκριθούμε, γιατί ε, δυστυχώς καταστράφηκαν υποδομές, στέγη, καλλιέργειες και γι' αυτό χρειάζονται πολύ υψηλά κονδύλια. Το Πακιστάν δεν μπορεί να ανταποκριθεί από μόνο του. Ξέρετε ότι καταπολεμούμε την τρομοκρατία τα τελευταία δύο με τέσσερα χρόνια για τις ανάγκες αυτού του πολέμου χάσαμε 42 με 50 ε, δις δολάρια και βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις επιθέσεις στα οικονομικά μας κέντρα. Ε, αντιμετωπίζουμε μία ε, δεινή οικονομική κατάσταση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Χαίρομαι που ακούστηκε μία φωνή σήμερα το απόγευμα σε σχέση με την αρρωγή αλλά και πέραν αυτής της άμεσης αρρωγής, διότι μιλάμε για τη φάση ανοικοδόμησης όπου χρειάζονται επιπρόσθετα δις δολάρια και με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και των ε, χρηματοδοτικών οργανισμών θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά την πρόσβαση στις αγορές. Όπως σας είπα, τα μέσα μας είναι περιορισμένα και έχουμε περιορισμένες δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Πακιστάν έτσι ώστε να έχει ευρίαση, ευρία πρόσβαση, με συγχωρείτε, στην αγορά για να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να ανταποκριθούμε σε αυτή την μεγάλη καταστροφή. Σας ευχαριστώ για την άμεση αρρωγή και βοήθειά σας γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αντουάν Κρεράρ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Επίτροπε, γιατί ε, μας είπατε ποια ήταν η αντίδρασή σας και η άποψή σας αφού είδατε την κατάσταση επιτοπίως. Αντέδρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Τονίσατε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα, διότι δεν μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια μόνο στο βορρά που υπάρχει μεγάλη σύραξη, αλλά και στο νότο που ζει αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Τώρα μιλάμε για την ε, πρωτογενή ανάκαμψη και σας υποστηρίζω σε αυτό. Ζητήθηκαν 537 εκατομμύρια και θα, θα υπάρξει και μία νέα έκκληση στις 17 Σεπτεμβρίου. Η δέσμευση αυτή υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών μελών έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε μόνο την, το ανθρωπιστικό σκέλος αλλά και το σκέλος της ανάκαμψης. Θα ήθελα να συζητήσουμε και την ε, εφοδιαστική, μάλλον την επιμελητιακή βοήθεια, γιατί εδώ υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, χρειάζονται ελικόπτερα σε αυτή τη χώρα. Η χρηματοδότηση μπορεί να επιτρέψει την ύπαρξη αυτών των ελικοπτέρων και οι δωρητές θα έπρεπε να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα ελικοπτέρων για πολιτικούς σκοπούς έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόσβασιμότητα του, του λαού. Με συγχωρείτε γιατί έχετε υπερβεί το, το χρόνο σας. Ε, ο κύριος Καρτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα ήθελα να μας απασχολήσει η κατάσταση στο Πακιστάν, ιδιαίτερα ως προς τα παιδιά. Υπάρχουν 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών που έχουν πληγεί άμεσα από αυτή την καταστροφή. Πρόκειται για μια ευάλωτη, την πιο ευάλωτη κατηγορία σε όλες τις ε, παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχει ε, διάρρεια, υπάρχει χολέρα, υπάρχουν πολλές αιστείες και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρξουν ε, παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, της υγιεινής και της, ε, των διατροφικών αναγκών. Επίσης μιλήσατε και για την κατάσταση των γυναικών. Τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετικές ανάγκες. Θα πρέπει να προβούμε στη σωστή στοχοθέτηση των παρεμβάσεών μας. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι η χρηματοδότηση είναι ύψη τη σημασία το ένα 50% για να ανταποκριθούμε στο 50% των αναγκών χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Ευχαριστώ κύριο Σίμω Μηθυρή από την, ε, το Διεθνή Ρηθρό Σταυρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Έχω τέσσερα σημεία τα οποία έχω σημειώσει να αναφέρω. Πρώτον, συμφωνούμε απολύτω για τα θέματα τη ανθρωπιστική καταστροφή. Είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή μεγαλύτερη από ότι ο σεισμό στο Πακιστάν το 2005 και από το τσουνάμι στην Ασία το 2005 ε, και ε, επίσης ε, σε σχέση με το σεισμό στην Αιτή επίσης είναι μεγάλη καταστροφή. Όπως ανέφερε και η Επιτροπή, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η Ερυθρέα η Έλληνο, ε, είναι εγκαταστημένη τόπου και προσπαθούν να ε, συντονιστούμε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες σε όλα τα μέρη της χώρας η ανταπόκριση ήταν αργή, μόνο κατά 50% καλύπτουμε αυτή τη στιγμή τα αιτήματα και υπάρχει ε, αίτημα για περισσότερα χρήματα τα οποία προς το παρόν δεν έχουν διατεθεί. Άρα ε, έχουμε ε, πρόβλημα και βασιζόμαστε στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ανασυγκρότηση, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ορίζοντα πενταετίας μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φωνσουά Μπελάν, Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ο Ερυθρός Σταυρός αναθεώρησε, ε, ε, επανεξέταση όλη την κατάσταση στην αρχή τη της καταστροφής αυτής και προσπαθούμε μαζί με τις αρχές του Πακιστάν να συνδυάσουμε τις προσπάθειε μα με τις προσπάθειε ε, της Ερυθράς ημισελήνου. Ε, καταφέραμε να στείλουμε ε, και επιστηστική βοήθεια και μη επιστηστική βοήθεια που έφτασε σε ε, πάνω από 300.000 άτομα. Και τώρα σε μετά από τα πρώτα 57.000 ελβετικά φράγκα που είχαμε στείλει, στείλαμε άλλα 134.000 ελβετικά φράγκα συνολικά. Στέλνουμε συνδρομή και σε τρόφιμα και σε άλλα είδη εκτός από τρόφιμα. Ε, και ελπίζουμε να φτάσουμε να καλύψουμε περίπου 700.000 άτομα με τη βοήθεια αυτή. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το θέμα της ασφάλειας. Σε πολλές περιοχές, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σύραξη και ε, ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το έργο, ε, αυτών, ε, το έργο αυτών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και σίγουρα η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι πολύ χρήσιμη. Η κυρία Καθήν Σίκ από το Voice. Το Voice είναι μία από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τα σχόλιά μα. Η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ε, όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, έχει σημασία ε, και το ποσό που θα δοθεί, αλλά και οι δεσμεύσει που θα δοθούν. Ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν δώσει τη δέσμευσή του, ε, που όμω δεν τηρείται πάντοτε. Και η ευελιξία όσον αφορά τα κονδύλια είναι πολύ σημαντική για να μπορούμε να προωθήσουμε την ανασυγκρότηση και για να μπορέσει να υπάρχει υπάρξει αποκατάσταση ε, των ε, ζημιών των πλημμυρών. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά καθυστερούν πάρα πολύ τα κονδύλια. Και αυτό δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει σχέση με τα κράτη-μέλη και έχει σχέση με τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δρούν σε τέλη των ΗΕ. Το Πακιστάν έχει δραματικές εμπειρίες από αυτό και στο παρελθόν και είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε την κατάσταση για να μπορέσουν όλοι να δουλέψουν καλύτερα. Η διαφοροποίηση της χρηματοδότησης επίσης είναι σημαντικό χρειαζόμαστε χρηματοδότηση προς όλους και προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και προς ε, ε, όλους και τα Ηνωμένα Έθνη και όλους όσους ε, δρούν επί τόπου. Ε, επίσης βοήθεια προς τα παιδιά και εκπαίδευση που πρέπει να παρασχεθεί επιγόντως. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα, έχετε το λόγο για να κάνετε τις τελικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και για την υποστήριξη προς εμένα και το επιτελείο μου. Θα ομαδοποιήσω κάπως ε, τις απαντήσεις μου. Τρία είναι τα βασικά ζητήματα. Πρώτον, για τη χρηματοδότηση, πώς ε, οργανώνουμε την ανταπόκριση, ποια ζητήματα πρέπει να ε, χειριστούμε σε σχέση με τη μελλοντική ανοικοδόμηση, την οικονομική πτυχή κυρίως. Δεύτερον, ανάπτυξη, δημοκρατία, εξτρεμισμός, τι επίκειται, τι, τι, μέλ, τι μέλ γενέστε μετά τις πλημμύρες και τρίτον συντονισμός, προβολή της δράσης μας, ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από το παρελθόν και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις μελλοντικές προσπάθειες παρέμβασης. Για τη χρηματοδότηση πρώτα απ' όλα. Ε, πολύ αναφέρθηκαν στο ότι χρειάζεται να συλλεχθούν κονδύλια όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου και ένα συγκεκριμένο ερώτημα άκουσα. Ε, με ρωτήσατε από η Κίνα, η Ινδία και είπα τι έχουν δώσει. 50 εκατομμύρια δολάρια είναι η δέσμευση των ΗΠΑ και ενδέχεται να την αυξήσουν από ό,τι καταλάβαμε. Η Ινδία 5 εκατομμύρια, η Κίνα ε, μικρότερο είναι το κονδύλι της προς το παρόν και δίκιο έχουν οι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συλλογή κονδυλίων, αλλά υπάρχει καλή συμφωνία αυτή τη στιγμή, διότι αλληλέγγυα έχουμε επικουρήσει το Πακιστάν ε, και ενεργώς έχουμε ζητήσει βοήθεια και από άλλους δωρητές. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε ισχυρότερη στήριξη από διάφορες άλλες χώρες. Ένα δισεκατομμύριο είναι συνολική βοήθεια, αλλά εξαρτάται γιατί ε, ε, δεν ξέρουμε ακριβώς ε, αν πρόκειται για την ανοικοδόμηση ή για την, την άμεση ανακούφιση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια, να ξέρουμε πού πάνε τα κονδύλια. 900 εκατομμύρια δολάρια θα έρθουν από την ε, ε, τράπεζα, την Ασιατική ε, Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επίσης υπάρχουν συζητήσεις με τον Επίτροπο Πίμπαλξ, ώστε ενδεχομένω να αυξήσουμε και τα κονδυλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη δεν έχει περατωθεί η συμφωνία. Πάντως είναι ήδη σαφές πως το Πακιστάν και ευχαριστώ που το αναφέρατε. Το Πακιστάν επιμένει για τα εμπορικά ζητήματα. Ε, μία οδός είναι η βοήθεια, άλλη οδός για να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα είναι το εμπόριο, ε, το άνοιγμα των αγορών μας. Όπως είπα και στις πακιστανικές ε, αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κάνει πολλά πράγματα για να ανοίξει ε, τις αγορές της για τα πακιστανικά προϊόντα. Είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός ε, του Πακιστάν. 20% περίπου των προϊόντων περνούν ατελώς. 60% ε, την χάνουν, διάφορες, την χάνουν διάφορων δοσμολογικών μειώσεων. Οπότε σωστή είναι η προσέγγιση των Πακιστανικών αρχών να προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συζητούν την, το περαιτέρω ανοίγμα των αγορών θα, όπως είπα και στις πασικιστανικές αρχές, είναι πολύ απλό. Στον εμπορικό τομέα χρειάζονται δύο για να γίνει ο χορός. Η Ευρώπη προφανώς είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Είμαστε δημοκρατικοί ακόμη και σε εμπορικά ζητήματα και πάντοτε τα θα υπέρ της φελευθεροποίησης του εμπορίου. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πληρούνται και κάποιοι όροι ε, από το Πακιστάν. Δηλαδή για ζητήματα που είναι ήδη επιτάπητο. Σας επιστρέψει στις ε, συζητήσεις ε, που, τις προϊούσες συζητήσεις να δει τι περαιτέρω προσπάθειες μπορεί να κάνει. Ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, σε σχέση με το Πακιστάν επηρεάζει τις σχέσεις της και με άλλους εμπορικούς εταίρους. Όντως είναι σε κατάσταση ανάγκη στο Πακιστάν και πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, αλλά θα πρέπει να είμαστε και συνεπείς. Και είπαμε, ο και ο Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν καλωσόρισαν ε, τα σχόλιά μου σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και τους προσκαλέσαμε και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, δεν είμαι σίγουρη ότι δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση για το χρέος. Ε, πάντως, όταν βαρύνεται έτσι μία χώρα, γίνονται διάφορες συνδυασμένες προσπάθειες για να ορθοποδήσει η χώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων και για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση θα καλύψουμε όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες για να ενισχύσουμε την ανοικοδόμηση. Και όπως ε, είπαν ε, τα μέλη της Επιτροπής, υπάρχει το θέμα ε, της ανοικοδόμησης, ναι μένα, αλλά Υπάρχει και το θέμα της αναδιοργάνωσης των θεσμών, ε, όπως και στην ΑΕΤ. Δηλαδή, αν έχετε τα χρήματα, αλλά δεν έχετε τους φορείς, τους θεσμούς, δεν μπορούν να διοχετευτούν τα κονδύλια. Επίσης, ε, για τη διαχείριση των καταστροφών πρέπει να ενισχυθούν οι θεσμοί, σας είπα ότι υπάρχει μία ε, επιτροπή, 23 άτομα δηλαδή, για να συντονίσουν όλες τις προσπάθειες. Εγώ έχω ένα επιτελείο 54 ανθρώπων για να συντονίσω τη δράση των κρατών μελών. Και όταν είδα τον επικεφαλής ε, του Πακιστάν με αυτή την πελώρια καταστροφή στα χέρια του και με αυτή την ε, μικρή ομάδα των 23 μελών να προσπαθεί να συντονίσει την καταστροφή, Τορυβήθηκα. Για, τις, ε, για την ανταποκρισιμότητα στις κλιματικές αλλαγές, το climate resilience. Ε, είδαμε τα τελευταία χρόνια στις υπηρεσίες μας ότι υπαρίσταται ανάγκη ανθρωπιστική πόροι να διοχετεύονται και για την αύξηση της ε, ανταποκρισιμότητας. Το 10% του προϋπολογισμού μας εκεί πάει. Για να προετοιμαστούμε έχουμε τον Τύπακ, Δηλαδή δράσεις που βοηθούν τις χώρες ώστε να είναι λιγότερο ευπαθείς. Δηλαδή, άμα έχουν μικρότερες ανάγκες επιλυγής σε χώρες, ε, φυσικά χρειάζεται και λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Και πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας ε, στο μέλλον ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε υψηλές φιλοδοξίες σχετικά με αυτό. Για τη δημοκρατία και τον εξτρεμισμό, περνώ στο δεύτερο θέμα διάφορα μέλη της Επιτροπής σχολίασαν το ζήτημα αυτό. Προφανώ η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είναι αμερόληπτη πολιτικός πώς ε, οφείλουμε να είμαστε ουδέτεροι. Είναι σημαντικό να ξέρουμε βέβαια αν βελτιώνεται ή επιδεινώνεται η κατάσταση της ασφαλείας, ε, γιατί επηρεάζει και την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όταν ήμουν εκεί, ε, ρώτησα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις τι πιστεύουν, Εάν δηλαδή έχουν απτά τεκμήρια πώς χρησιμοποιούνται οι πλημμύρες από τους εξτρεμιστές Ε, ως πρόσχημα, αν τις εκμεταλλεύονται. Από ό,τι κατάλαβα από τις απαντήσεις, ε, δεν πρόκειται για ε, γενικευμένο πρόβλημα. Δεν νομίζω να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις, αλλά σίγουρα μέσα στο χάος θα γίνουν, θα υπάρξουν απόπειρες να επηρεαστούν οι πεπιθήσεις των ανθρώπων οι πακιστανικές αρχές αφώς μου είπαν ότι όλοι ζητούν τη βοήθεια. Εάν υπάρχει βοήθεια, ε, κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσει κατά του εξτρεμισμού και υπέρ της δημοκρατίας. Κυρίως ε, αν θεσπίσουμε μέτρα για διαφάνεια και λογοδοσία, όχι μόνο για τα, τους δικούς μας τους πόρους, αλλά και για τους, για τους πακιστανικούς πόρους. Και το αντίστροφο ισχύει. Εάν δεν βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αν είναι ε, σε απόγνωση, αν υπάρχει χάος, τότε ενδέχεται να υπάρξει και ε, αποσταθεροποίηση, ελοχεύει ο κίνδυνος. Είναι ένα ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Για τις γυναίκες πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να απαντήσω. Εγώ εντυπωσιάστηκα ε, σε αυτή την περιοχή που επισκέφθηκα, που είναι μάλλον συντηρητική. έχουν καταστραφεί όλα σε αντίσκηνα μένει ο κόσμος και ε, ε, οι γυναίκες μένουν μέσα στους ε, καταβλισμούς και οι άντρες είναι απ' έξω. Φυσικά υπάρχουν υγειονομικά προβλήματα. και πολλά νοικοκυριά σίγουρα δεν τα αναλαμβάνουν οι γυναίκες γιατί είναι συντηρητική περιοχή όπως σας είπα. Τώρα, ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, πάμε τα κορίτσια στο σχολείο ή τα σχολεία στα κορίτσια, όπως θέλετε να το δείτε πολιτικά. Θα πρέπει να διοχετεύουμε τα κονδύλια στα νοικοκυριά που είναι επικεφαλής οι γυναίκες. Εκεί ε, κλείνοντας αυτό το θέμα θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Σε σχέση τώρα με τα βιώματά μας στην ΑΕΤ, τι έχουμε μάθει. Χρειάζεται η Ένωση ισχυρότερο μηχανισμό συντονισμού των δράσεών μας, με το που ενεργοποιεί το μηχανισμός, ε, οδηγεί σε μια συνεκτική ε, αντίδραση. Αλλά ε, ε, δεν είναι υποχρεωτική αυτή η συνέπεια που δείχνουμε. Εξαρτάται από την καλή θέληση όλων. Εάν όμως έχουμε ε, πόρους ε, που θα είναι στη διάθεσή μας θα τα καταφέρουμε καλύτερα στο μέλλον. Δηλαδή ε, εγώ από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι αντιδρούν πολύ γρήγορα τα κράτη-μέλη όταν του ζητείτε η βοήθεια, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω, ε, εναγωνίως περιμένω να δω σε ποιο βαθμό θα βοηθήσουν άλλες χώρες. Ε, και Από ό,τι βλέπω, από τα μέσα που προτίθεται να διαθέσουν τα κράτη-μέλη, μπορούμε να αντιδράσουμε ταχαίως και με συντονισμένο τρόπο. Διότι όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνδυάζουμε ε, τα, ε, τις, ε, τη βούληση των 27 κρατών μελών Ε, και ξέρουμε ότι δεν συμφωνούν ε, όλες οι χώρες ανάλογα με το αν έχουν πληγεί και οι ίδιες στο παρελθόν. Ας κάνω και λίγη αυτοκριτική. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένε φορέ προβάλλει το δικό της το έργο και δεν αναφέρει επαρκώ ότι πρόκειται για συνδυασμένη προσπάθεια 27 κρατών μέλων. Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει προ όφελο των πολιτών. Θα πρέπει όλοι να μιλάμε με μία φωνή. Και Τώρα για τα, ε, το στρατιωτικό εξοπλισμό και του στρατιωτικού πόρους, ναι, έχουν κυρία σημασία ενίοτε όπως στην ΑΕΤ. Ε, Παραδείγματο χάρη, αεροσκάφη για να πηγαίνει η βοήθεια των κρατών μελών στο Πακιστάν χρησιμοποιήθηκαν, αλλά είναι και ευαίσθητο το ζήτημα και ε, μπορεί να κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, εκτό και αν υπάρχει ο σωστό συντονισμό. Μα τι σημαίνει επιτέλου σωστό ε, συντονισμό. και το ίδιο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κοινέ προσπάθειες. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Εάν θεωρείτε ότι δεν είναι καλή ιδέα η στρατιωτική βοήθεια, θα σας ακούσουμε. Ε, γιατί έτσι θα έχουμε το ευρύτερο δυνατό πεδίο δράσης και παρέμβασης. Ε, ένα βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής μας ε, ε, πολιτικής είναι να προβάλλουμε με ποιο τρόπο συνδυάζουμε και διαθέτουμε τους πόρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μπορούμε να αντλήσουμε πολλά περισσότερα διδάγματα και από την ΑΕΤ και από το Πακιστάν για την ΑΕΤ. Ένα σημείο θα ήθελα να αναφέρω για το ανθρωπιστικό κομμάτι. Είχαμε πολύ καλές επιδόσεις. ανησυχούσαμε ε, ότι θα ε, εξαπλωθούν επιδημίες, δεν έγινε αυτό. Ε, φοβούμασταν το χάος, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Όταν φτάνουμε στην ανοικοδόμηση όμως, όπου έχουν προεξάρχουσα σημασία τα θεσμικά ζητήματα, τότε βλέπουμε τα πραγματικά προβλήματα, γιατί έχουμε ε, πολύ υψηλά κονδύλια, αλλά πολύ ισχνό ε, θεσμικό μηχανισμό για την απορρόφησή τους. Και γι' αυτό σας λέω ότι στο Πακιστάν πρέπει να φροντίσουμε και τις δύο πλευρές για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο στάδιο της ανοικοδόμησης. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που κάνατε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ σήμερα. Eh bien voilà, Madame Jolie était en partie un peu plus tôt. Η κυρία Ζολή χρειάστηκε να φύγει λίγο νωρίτερα. Κλείνουμε λοιπόν αυτή τη συνεδρία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο και να ευχαριστήσω και όλου εκείνου που έλαβαν το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την ιδιαίτερα σημαντική συνεδρία. Θα τα πούμε σύντομα.